Diamo inizio alla nostra commissione. Συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Έχουμε μεταξύ μας ε, τον Σουηδό Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριο Εσκίλ Έρλανσον. Σε ευχαριστούμε Εσκίλ που βρίσκεσαι σήμερα ανάμεσά μας και προβλέπεται μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πρόγραμμα της Σουηδικής Προεδρίας. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν προβλέπεται η ομιλία του ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου, κ. Έσλαντσον και μετά θα ακολουθεί συζήτηση και θα περάσουμε στην στις ε, έρωτα ε, Έχουμε μία ώρα καιρό μπροστά μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι αγαπητά μέλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής σας για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας όσον αφορά τη γεωργία και την αλία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό το οποίο έχει, πιστεύω, ε, για μας μια ιδιαιτερότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε ως Σουηδική Προεδρία ένα νεοεκλεγέν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως ε, είμαι περίεργος και αναμένω με ανυπομονησία το μήνυμα το οποίο θα περάσει από εσά προ τα εμένα στην νέα μου αυτή ιδιότητα ω Προεδρεύον του Συμβουλίου. Θα πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία μας αυτό το φθινόπωρο θα είναι λίαν επιτυχής. Η Σουηδική Προεδρία έχει τρεις βασικές προτεραιότητες υπό την ε, δική μου, ε, υπό τον δικό μου τομέα ευθύνη. Και τρει βασίζονται στη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρί κατάχρηση. Οι τρεις προτεραιότητες είναι η μακροπρόθεσμη αηφόρος ε, αλία, τρόφιμα και κλίμα σε προκλήσεις και η σωστή κτηνοτροφία με υγιή ζώα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσω την προσοχή μου σε αυτούς τους τρεις τομέας και, ε, τομείς και να σας παρουσιάσω ε, την κατάσταση γενικά όσον αφορά τα τρόφιμα, το κλίμα και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η εξασφάλιση ε, η του της επάρκειας τροφίμων είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση δεδομένου ότι ο πληθυσμός της γης θα φτάσει περίπου τα 9 δισεκατομμύρια το 2050 και μαζί με άλλα πολυμερή, άλλους πολυμερείς οργανισμούς, τον ΦΑΟ, ε, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Ε, η συνεργασία μας θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση ε, της σύντησης όλου του πληθυσμού του, της υφηλίου και ε, γι' αυτό αυτό το φθινόπωρο ε, το ε, Συμβούλιο του ΦΑΟ το οποίο είναι γνωστό υπό τον τίτλο Conference θα συνέλθει για να συζητήσει αυτά τα, θέματα. Η Προεδρία θα μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα, θα προσπαθήσει να δώσει μια νέα όθηση στις εργασίες του ΦΑΟ προς αυτή την κατεύθυνση της επάρκειας τροφίμων. Μία άλλη παγκόσμια πρόκληση είναι βεβαίω το κλίμα. Το κλίμα. Η γεωργία παίζει ένα ρόλο κλειδί στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά πρέπει επίσης να προσαρμοστούμε στις αλλαγές που αντιμετωπίζουμε ε, και ιδιαίτερα στην αλλαγή των συνθήκων ε, επάρκειας ύδατος και στις νέες ε, επιζωοτίες, στις αρρώστιες των ζώων και των φυτών και ο γεωργικός τομέας είναι μέρος του προβλήματος αλλά και μέρος της λύσης για μία αηφόρο ε, παραγωγή ενέργειας. Την, ε, στην πρώτο, πρώτο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας ε, υπό την Σουηδική Προεδρία τον Ιούλιο οι Υπουργοί συζήτησαν την προσαρμογή της γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί στην Υπουργική Συνάντηση στο Βέξιο ε, και θα συζητήσουμε τα θέματα της γεωργίας και του κλίματος και επίσης ε, το θέμα της ε, μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ελπίζω ο πρόεδρο τη Επιτροπή, ο Σπάλο θα μπορέσει να έρθει στο Βέξιο και να, για να συμβάλλει σημαντικά σε αυτέ τι συζητήσει. Ε, πάλι στον τομέα των, του κλίματος και των κλιματικών ε, αλλαγών θα οργανώσουμε δύο περαιτέρω συνεδριάσεις στη Σουηδία το φθινόπωρο. Η μία θα έχει τον τίτλο «Κλίμα, έξυπνα τρόφιμα, Climate Smart Food» και θα συζητήσουμε τι μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί τροφίμων και οι καταναλωτές για να μειώσουν τις επιπτώσεις του, στο, της παραγωγής τροφίμων στο, στο κλίμα, στις κλιματολογικές συνθήκες η άλλη διάσκεψη θα έχει επικεντρωθεί στην έρευνα ε, και βασικά στην έρευνα ε, που θα καλύπτει τις υπαίθριες περιοχές και θα βοηθήσει τις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις νέες αλλαγές του κλίματος. Αυτές, αυτές οι δύο συνεδριάσεις θα συζητήσουν επίσης και το θέμα της ε, αηφόρου παραγωγής βιοενέργειας. Η Γαλλική Προεδρία έχει αρχίσει τη συζήτηση τότε για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής και η ε, Προεδρία της ε, Δημοκρατίας της Τσεχίας τη συνέχισε στην ε, συνάντηση που έγινε του Συμβουλίου τον που θα γίνει τον Οκτώβριο, θα κάνουμε μια συζήτηση γενικά της πολιτικής για το μέλλον της, του γεωργικού τομέα με επίκεντρο την ανάπτυξη της υπαίθρου στον, ε, ε, οι διαβουλεύσεις που γίνονται στον ΠΟΕ είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον και η Προεδρία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ελπίζει να καταλήξει γρήγορα ο γύρος της Ντόχα. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί καθημερινά είναι το ρυθμιστικό σύστημα και δεν θέλουμε να είναι υπερβολικά βαρύ έτσι ώστε να δημιουργεί προσκόμματα στις ενεργές μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν απλοποίηση. Είναι βέβαια εύκολο να μιλάμε για απλοποίηση, αλλά πολύ δύσκολη η εφαρμογή της. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η σημασία η σημασία που έχει ε, να βρεθούν οι παραγωγοί και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι του τομέα στο επίκεντρο των συζητήσεων θα ξεκινήσουμε ε, τη συζήτηση αυτού του θέματος γενικά με, την, ε, με, με, με, με πρώτο θέμα τη μείωση του διοικητικού άχθους, του διοικητικού βάρους και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε μια ταχύτερη λειτουργία του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην καθημερινή ζωή και μια απλοποίηση των κανονισμών θα γίνει Συμβούλιο ε, Υπουργών τον ε, Νοέμβριο όπου θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και η Κομισιόν θα παρουσιάσει εκεί τις προτάσεις της. Οι προτάσεις αυτές θα βασίζονται στο, στις 39 συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες υιοθέτησε το, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στη συνάντηση του Μαΐου. Ελπίζω να έχουμε να συνεχιστεί η στενή και καρποφόρα συνεργασία μαζί σας σε αυτόν τον τομέα. Διαφορετικά θα κολλήσουμε ε, και θα κατακλειστούμε από μια χιονοστιβάδα ε, ε, χαρτιών και φακέλων που θα μας εμποδίσει την πρόοδο του θέματος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην Προεδρία μας θα είναι η αντιμετώπιση βεβαίως οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία έχει πειράσει όλους τους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε αυτή αυτό το γεγονό να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ιδιαίτερα εν ώψη της κρίσης στην αγορά του γάλακτος. Οι τιμές του γάλακτος έχουν, πέσει ταχύτερα τους τελευταίους 12 μήνες από ό,τι μπόρεσε κανείς να προβλέψει. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με κατόπιν ετήσεώ του, η Κομισιό παρουσίασε μια ανάλυση του γαλακτοκομικού τομέα στο τέλο Ιουλίου και είναι στην πρώτη σειρά προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και έτσι το Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα το ταχύτερο να συζητήσει υπό τη Σουηδική Προεδρία το Σεπτέμβριο αυτό το θέμα, ε, το, την ερχόμενη Δευτέρα μάλιστα. Και τον Ιούλιο η Κομισιόν είχε παρουσιάσει την πρόταση για μια ε, εκτεταμένη περίοδο παρέμβασης για τα προϊόντα γάλακτος και και λόγω αυτής της πρότασης της Κομισιόν για την παράταση της περίοδου παρέμβασης η Προεδρία πιστεύει ότι ένα άλλο θέμα υψής της προτεραιότητας είναι η λήψη απόφασης το ταχύτερο δυνατόν. Γι' αυτό ε, το Συμβούλιο υπάρχει ευρία υποστήριξη σε αυτή την πρόταση αλλά εξαρτώμαστε και από εσά. Το Κοινοβούλιο και την ε, έξεση σας, τη γνωμοδότησή σας να την έχουμε στα χέρια μας το ταχύτερο δυνατόν. Θα ήθελα τώρα να, γυρίσω στα, ε, να επανέλθω στα μέτρα τα οποία ε, ε, στοχεύουν στην ενίσχυση του Flect, που είναι το πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τα δάση τη διαχείριση των δασών και την εμπορία δασικών προϊόντων. Πέρσι τον Οκτώβριο η Κομισιόν είχε προτείνει ε, την υποχρέωση των ε, εμπορευομένων, του τομέα που, που δημιουργούν, παράγουν και διαθέτουν ξύλινα προϊόντα, προϊόντα ξυλία στην αγορά, να τηρούν ορισμένους κανονισμούς, ορισμένες προδιαγραφές. Αυτό είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει πάρα πολλούς διαφορετικούς κλάδους του τομέα της εμπορίας και παραγωγής προϊόντων ξυλίας και θα το εξετάσουμε και αυτό με μεγάλη προσοχή στο Συμβούλιο προς το τέλος του φθινοπόρου. Η τρίτη προτεραιότητα που σας είπα προηγουμένως είναι η σωστή κτηνοτροφία με υγιή ζώα. Είμαι πεπισμένος ότι μια σωστή κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να είναι υγιή τα ζώα. Θα κάνουμε ένα, ε, συνέδριο τον Οκτώβριο το οποίο θα αφοσιωθεί σε αυτό το θέμα και ελπίζω εδώ να παίξετε ένα πολύ ε, δημιουργικό ρόλο εσεί του, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα οργανώσω και ένα γεύμα μεσημεριανό για να συζητήσουμε το θέμα της υγιού εκτροφή ζώων και των υγιών ζώων το φθινόπωρο. Υπάρχουν πολλά άλλες προτάσεις στο τραπέζι που έχουν σχέση με την ε, ε, ε, ευζοία των ζώων. Ένα από αυτό είναι, μία από αυτές προτάσεις είναι η πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της νομοθεσίας την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Θα συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο για να δούμε αν είναι δυνατόν να επιτύχουμε μια συμφωνία σε αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια του, της συναπόφασης της διαδικασίας Βέβαια, θα θέλαμε πάρα πολύ να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτές με την νομική ε, βάση ε, προς το τέλος του φθινοπόρου. Επίσης, έχουμε πρόθεση να συζητήσουμε ε, με τη συνεργασία της Κομισιόν κατόπιν της ανακοινώσεώς της το πρόγραμμα δράσης για την προστασία και ευζοία των ζώων. Όσον αφορά τώρα τον τομέα της υγείας των ζώων, η Προεδρία έχει δεσμευθεί να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγείας Ζώων. Εδώ ε, ε, προχωρούμε με, με, γρήγορα βήματα στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις νομοθετικές προτάσεις το 2010. Η υγεία ε, των ζώων και η πολιτική προστασία τους πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στι απαιτήσει τη σύγχρονη εκτροφής και τη σύγχρονη ε, κτηνοτροφής εν ώψη δε των νέων κινδύνων και αρρωστιών που ε, σημειώνονται στον τομέα. Ε, επίσης πρέπει να απλουστεύσουμε την νομοθεσία σε αυτό τον τομέα έτσι ώστε να μπορέσουν και οι παραγωγοί του, στον τομέα αυτό να προσαρμοστούν χωρίς επιπλέον διοικητικό φόρτο για την ε, ζωική υγεία, ε, μετά από την υγεία των ζώων, θα ήθελα να προχωρήσω σε θέματα τροφίμων. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι εξαιρετικά σημαντική για τους καταναλωτές και πρέπει να βρούμε μια ε, καλή ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην πρόταση αυτή η οποία αφορά την, προμήθεια, την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα και ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να καταλήξουμε σε ένα κονσένσους μέσα στο Συμβούλιο το φθινόπωρο. Όσον αφορά τώρα τα λεγόμενα νέα τρόφιμα, novel foods, εδώ θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την πολύ καλή εργασία που έκανε η προηγούμενη Προεδρία της ε, Τσεχίας για να προετοιμάσουμε τη δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Καταλήγοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα εργαστούμε για την καλή εφαρμογή της συνθήκης ε, της Λισαβόνας εάν τεθεί ενισχύ το φθινόπωρο. Η συνθήκη της Λισαβόνας θα φέρει μεγάλες αλλαγές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δι στον τομέα της γεωργίας. Η εφαρμογή της συνθήκης λοιπόν πιστεύω ότι θα μας ε, διευκολύνει στο να προχωρήσουμε γρήγορα και με πιο αποφασιστικά βήματα. Αυτή, αυτή φίλη μου ήταν μια ε, σύντομη ενημέρωση για τις προτεραιότητες Τη της προεδρία και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει και σχόλια. Σα ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας έκανες, κάτι το οποίο μας διευκολύνει στο να εξετάσουμε το πρόγραμμα της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Τώρα, κάνοντας αναφορά και στην συναπόφαση, θα ήθελα να τονίσω τις ευθύνε που φέρει η Επιτροπή μας ε, πάνω στο ζήτημα σήμερα, μιλώντας ε, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα θέλαμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει το Συμβούλιο τις προσεχείς εβδομάδες. Έχουν ζητήσει το λόγο πρώτα απ' όλα ο Άλμπερντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Έλανσον. Χαίρομαι που η Σουηδία έχει την Προεδρία του Συμβουλίου και άκουσα με ενδιαφέρον της, ε, την ενημέρωσή σας. Αναφέρετε την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Ρωτώ λοιπόν εάν κατά το χρονικό διάστημα της Σουηδικής Προεδρίας θα αναλυφθούν και άλλες πρωτοβουλίες παραδείγματο χάρη εκεί όπου υπάρχει εσφαλμένη ενημέρωση του καταναλωτή να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις και ε, επίσης αν θα προωθήσει το θέμα της βελτίωσης των ε, πληροφοριών που αναφέρονται στις ετικέτες των τροφίμων. Είπατε ότι η επάρκεια των τροφίμων πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους τους κατοίκους ε, της Ιφιλίου. Ε, σωστά βεβαίως, αλλά σε πολλές ε, τρίτες χώρες τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί είναι δημιουργία του ιδίου του κράτους. Παραδείγματος χάρη δείτε την περίπτωση της Ζιμπάμπουε ε, όπου πριν από μερικές δεκαετίες υπήρχε πλήρης επάρκεια τροφίμων και δύο εξαγωγές και τώρα οι άνθρωποι λιμοκτονούν ε, χωρίς να φταίνε, να φταίει κανείς άλλος για αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν θα λάβετε ορισμένα μέτρα ή τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε αυτή την κατάσταση. Είπατε επίσης ότι θα θέλετε να ολοκληρωθούν ε, ορισμένοι φάκελοι μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Α, ο, γύρος της Ντόχας στον ΠΟΕ. Θα ήθελα να ξέρω τώρα με, με ποιες, ε, υπό συνθήκες και με τι όρους ε, θέλετε να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα. Το θέμα είναι ότι ότι ε, αν επιτρέπουμε την εισαγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θα πρέπει να υφίστανται, να, να, να σέβονται, να υπάρχει συμμόρφωση στους ίδιους κανονισμούς όπως και στα δικά μας ε, τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσετε πολύ στενά τα στάνταρτ, τα πρότυπα αυτά βάσει των οποίων τα προϊόντα ε, παράγονται, παραδείγματος χάρη στη Βραζιλία, ε, εξάγονται και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε αφενό να μην παραβιάζουν τους δικούς μας κανονισμούς ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και αφετέρου να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που προσδίδεται ε, μεγάλη σημασία στην συζήτηση του μέλλοντος της γεωργίας και δόξα τω Θεώ ε, τα, θέματα είναι σοβαρά και δεν χρειάζεται πλέον να συζητούμε ε, αν θα τετραγωνίσουμε τα καρπούζια ή την καμπύλη των αγκουριών όπως είπε ο ομιλητής. Λοιπόν, ε, στις 12 ε, Μαρτίου μετά από την δήλωση της Επιτρόπου είχαμε, είχε ελεχθεί και είχε καταγραφεί στα πρακτικά για το γαλακτοκοπικό τομέα ότι έτσι όπως πηγαίνουν τα παράγματα τότε την Άνοιξη ο τομέας αυτός θα καταστραφεί ολοσχερός και θα επέλθει η πλήρης ισο, ισοπαίδωση των παραγωγών με τις τιμές αυτές του γάλακτος. Άρα και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Να σας ε, ευχηθώ το καλώς ορίσατε και εύχομαι στην χώρα σας, στη Σουηδία, καλή επιτυχία στο έργο της. Είμαι βέβαιος πως θα το πετύχει και μπόρεσα εξάλλου να εκτιμήσω τις ικανότητες της κυβερνήσεώς σας σε ό,τι αφορά την διαχείριση των κοινωτικών ζητημάτων στην προηγούμενη Προεδρία σας. Έχουμε κάποιες προκλήσεις βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες. Τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις ε, στον γαλακτοκομικού τομέα, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη και την επιβίωση πολλών γεωργικών, πολλών ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σας ε, ευχαριστώ που φροντίσατε να προτάξετε το Συμβούλιο Υπουργών στι 7 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που προτίθεστε να προωθήσετε και να υιοθετήσετε έτσι ώστε να παροτρύνετε την ε, λήψη των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να υποβάλει τα απαραίτητα μέτρα προς ε, εφαρμογή. Μέτρα που μέχρι, το παρόν, μέχρι τώρα μάλλον απαιτήθησαν ανεπαρκή θα ήθελα να παρατηρήσω πως τα μέτρα θα πρέπει να επεξαθούν και στο βούτυρο και στα τυροκομικά. Αυτό φυσικά θα επιλύσει τα προβλήματα, αλλά εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στην κοινή γνώμη. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψη της Προεδρίας επ' αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις, ε, που θα έλεγα ότι είναι μάλλον μεσοπρόθεσμες, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μελλοντικής ε, ΚΑΠ πιστεύω πως ε, μία από τις πρώτες δηλώσεις που κάνατε ως ε, Προεδρεύων δηλώσατε στο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πως η Σουηδία είναι υπέρ του περιορισμού των ενισχύσεων προς τους γεωργούς. Το, δεν θέλω να θίξω θέματα περί δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά γνωρίζουμε πως ο προπολισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μειώθηκε ενώ αυξήθηκε ο αριθμός ε, των ευεργετουμένων στον τομέα της ΚΑΠ. Πολλά από τα κριτήρια που κατανέμουν τις ε, ενισχύσεις τους γεωργούς είναι άδικα, αλλά το να δηλώνουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι ενισχύσεις προς τους γεωργούς σε μια στιγμή, σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη, καταλαβαίνετε πως ε, δεν μπορεί να με βρει σύμφωνο με αυτό το πολιτικό μήνυμα που θελήσατε να στείλετε. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα και σας εύχομαι εκ νέου καλή επιτυχία ως Προεδρία. Ο κύριος Νίκολσον ζήτησε το λόγο. James, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του, γιατί είναι δύσκολη καιρή που περνάει η γεωργία. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία, τουλάχιστον να και στον τομέα συγκεκριμένα και στον τομέα της αλίας, διότι πολύ, πολύ καιρό ασχολούμαι με αυτό και πρέπει να, κάτι να γίνει. Μιλήσατε για απλούστευση, κανονισμούς. Ε, ε, επίσημα όλα αυτά τα λέμε ε, γραφειοκρατία. Παρακολουθώ εδώ και καιρό τα θέματα αυτά. Όλοι μας λένε ότι θα εξαφανίσουμε την γραφειοκρατία, θα εξαφανίσουμε τη χαρτούρα και θα γίνουν πιο αποτελεσματικά τα πράγματα στη γεωργία. Όμως κάθε φορά που υποβάλλουμε μια καινούργια πρόταση δημιουργούμε περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Επομένως ρωτώ, εσείς γιατί δεν καταφέρετε καλύτερα από ό,τι οι άλλοι στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γεωργούς ε, ε, γιατί θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν συγκεκριμένη δουλειά τους, να παράγουν τροφές, να φροντίζουν τα ζώα τους και δεν θέλουν να έρθει κάποιος από το πανεπιστήμιο και να τους πει πώς να ε, διευθύνουν την εκμετάλλευσή τους, ε, το αγρόκτημά τους και ουσιαστικά δεν ξέρουν τίποτα που, που τους πάνε τα τέσσερα. Λοιπόν, εδώ στι Βρυξέλλε παράγουμε χαρτιά, παράγουμε πολλά χαρτιά και πρέπει να τα ε, περιορίσουμε κατά πολύ. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, τι γίνεται με αυτούς που εφαρμόζουν τους κανονισμούς που υιοθετούμε εδώ. Τους εφαρμόζουν σε τέτοιο τρόπο που δεν είναι ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη-μέλη και τελικά ε, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ε, ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Επομένως, εσείς και δεν τα καταφέρετε καλύτερα από τους άλλους. Πάντως σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα είμαι στο πλευρό σας. Ο άλλος στόχος είναι που συζητάμε αυτή την εβδομάδα είναι τι θα γίνει με, τους, με τον γαλακτοκομικό τομέα και ελπίζω ότι και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα, τα, θα το συζητήσουμε. Και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα αντιδράσει με τον, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον επίγοντα χαρακτήρα του προβλήματος. Τα αγροκτήματα εξαρτώνται από, την νομοθεσία αυτή και πολλοί αγρότες, πολλοί γεωργοί ε, από την περιοχή που προέρχομαι εγώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τον τομέα και δεν θα επιστρέψουν γιατί δεν τους συμφέρει. Ένα από τα πράγματα τα οποία λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε που ακούστηκε είναι η κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Έχετε υπόψη σας πώς αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση Εάν και εφόσον καταργήσουμε τι ποσοστώσει, η γαλακτοβιομηχανία θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Ε, άλλοι θέλουν να εξασφαλίσουμε μια ομαλή προσγείωση για τη γαλακτοβιομηχανία, έτσι όπως είχαμε πει και στο checklist. Ε, τελικά όμως ε, οι αποφάσεις που πήραμε όχι, δεν εξασφάλισαν, όχι δεν εξασφάλισαν ομαλή προσγείωση, ήταν από τις πιο ανώμαλες προσγειώσεις που έχουμε δει. Επομένως, μήπως μπορείτε να ξέρετε κι εσείς τι πρέπει να γίνει, να ξέρουμε κι εμείς θα πούμε στους ε, αγρότες μας ή θα πρέπει να επιστρέψουμε στο, στην αφετηρία να δεχτούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ε, τα φανταζόμασταν πριν από μερικά χρόνια και να επανεξετάσουμε τον, ε, τον όλο καταλακτοκομικό τομέα υπό το φως των όσων συμβαίνουν τώρα, λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμβαίνει και στις παγκόσμιες αγορές. Μάρτιν Όσλινγκ Ε, κύριε ε, ε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας εύχομαι κάθε τύχη, καλή τύχη και επιτυχία στις εργασίες σας, δεδομένου ότι λαμβάνετε, προεδρεύετε σε μια πολύ δύσκολη εποχή οικονομικής κρίσης και η γεωργία ε, υποφέρει πάρα πολύ. Πολλές φορές στο παρελθόν η Επιτροπή Γεωργίας ήταν ικανοποιημένη με τις απαντήσεις της ε, Κομισιόν πιστεύω ότι η γενική πρόθεση που επικρατεί είναι να περιμένουμε να τελειώσει αυτή η κρίση και χωρίς να, να λάβουμε κάποιες ριζοσπαστικές ενέργειες. Πολλοί λένε ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Έστω και αν το δεχτούμε αυτό όμως δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε διότι οπωσδήποτε δεν έχουμε βρει λύσεις. Το ότι να καθόμαστε ε, απραγείς και να περιμένουμε να περάσει πάνω το κεφάλι μας δεν είναι και η ιδανική λύση. Βεβαίως η, κρίση αυτή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιπτώσεις και σε άλλες ε, χώρες και αντίστροφα. Θα θέλαμε από εσά να ακούσουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Ε, το έχουμε πει ε, στον τομέα του γάλακτος ότι περιμένουμε με ανυπομονησία νέες πρωτοβουλίες να αναλυφθούν. Επίσης, Τι θα κάνετε με τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Θα συνεχίσετε την υπάρχουσα πολιτική ή θα... Ε, η πρόθεσή σας είναι να λάβετε περισσότερα μέτρα, πρόσθετα μέτρα και πιο αυστηρά για να ελέγχετε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων και των επιτρεπτών ε, ποσοστών ε, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στα εισαγόμενα τρόφιμα. Όσον αφορά τώρα το, το, το κλίμα, ναι, βεβαίως αυτό πρέπει να το συζητήσουμε γιατί πιέζουν και πάρα πολλές οργανώσεις περιβαλλοντικές. Ε, για το επισητιστικό τώρα θέμα για τα, τα τρόφιμα και την επάρκεια τροφίμων. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Γεωργίας προβάλλει τις, ε, τα αιτήματα των ε, τρίτων χωρών και δι των αναπτυσσόμενων χωρών ε, και τονίζουν ότι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο την επιβίωση των παραγωγών σε τρίτες χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες και την εξασφάλιση δικαίων εισοδημάτων, εισοδημάτων επιβίωσης στους ανθρώπους αυτούς. Τι θα κάνετε σε αυτό τον τομέα. η κυρία Γέγκερ. Δυστυχώ, δυστυχώς το μικρόφωνο της ναι, δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, χαίρομαι που ήρθατε σήμερα ε, ε, που μας παρουσιάσατε τις προθέσεις σας. Αλλά εγώ θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέμα της, του επισητισμού Τη υφηλίου. Από τη μία πλευρά πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των ε, τρίτων χωρών και από την άλλη πλευρά μας κατηγορούν ε, πολλές φορές ε, ότι εμείς δεν κάνουμε πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε τον επισητισμό των άλλων περιοχών του κόσμου. Ρωτώ λοιπόν πώς θα μπορέσουμε η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν πολύ καλά υψηλής ποιότητας εξού και ακριβά προϊόντα να και, αυτά γίνονται, αυτό γίνεται επειδή σέβονται και συμμορφώνονται ε, με τις ευρωπαϊκές συνθήκες ε, και παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. Πώς θα μπορέσουν λοιπόν να προσαρμόσουν τις τιμές τους ε, ώστε να μην διατίθεται τα προϊόντα αυτά σε τόσο υψηλές τιμές. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε με ευρύτατη ε, συνένεση και μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κάπολντο Σάντος, Κάπολας ε, εάν θα πολεμήσετε ε, για αυτήν την, τον προϋπολογισμό της Γεωργίας, Δηλαδή, εάν υπεραμεινθείτε των πιστώσεων για τη γεωργία με πάθος και ενεργητικότητα και να μην αφήσετε τα κονδύλια αυτά να διαραίουν προς άλλες κατευθύνσεις. Ε, πιστεύω ότι έχουμε ψηφίσει ένα ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο πολύ λογικό και ότι θα μπορέσετε να το υπερασπιστείτε αυτό. Επίσης, χαίρομαι που θα συνεχίσετε τις τι συζητήσει για την ευζοία των ζώων και για την προστασία των ζώων. Το είχαμε, αυτό, ε, είχαμε επιμείνει στη συζήτηση αυτού του θέματος και στην παλιά Επιτροπή Γεωργίας και θα επιμείνουμε και θα συνεργαστούμε μαζί σας και με την καινούργια Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικουλέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία σας και συμφωνώ με τα σχόλια που εξέφασαν οι συνάδελφοί μου, αλλά παράταση έχουμε και εγώ καλή επιτυχία. Έχω δύο θέματα που θα ήθελα να θίξω. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κομματιού της συνεδριάσεώς μας, το πρωί δηλαδή, ο Τσέχος Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβηκε η Τσεχική Προεδρία για τις ε, άμεσες ε, ενισχύσεις από το 2013. Ε, γνωρίζω πως η Σουηδία δεν συμφώνησε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο Μπρουνό και τα την μείωση των ε, επιδοτήσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν με ποιο τρόπο θα προχωρήσει η Σουηδική Προεδρία. Προτίθεστε να ξεκινήσετε ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη Δεύτερη ερώτηση. Ο Επίτροπο ε, εμφανίστηκε ενώπιον τη εμφανίστηκε ενώπιον τη Επιτροπή Προπολογισμών και πρότεινε κάποιες ε, πιστώσεις να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί ένα έλλειμμα 4,4 δισεκατομμυρίων στον τομέα του Γάρετ. θέλω να γνωρίζω εάν ε, έχετε υπόψη σας αυτή την πρόταση και αν κρίνετε αποδεκτή μια παρόμοια πρόταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Νικουλέσκου Λαβία. Κύριε Πρόεδρε και από πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διαθεσιμότητα που δείξατε προκειμένου να μας αναφέρετε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που προτίθεστε να προωθήσετε κατά διάρκεια της Προεδρίας ακούσαμε από πλευρά ε, συναδέλφων ε, να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε ένα τομέα, τον γαλακτοκομικό, που χαρακτηρίζεται σήμερα από σοβαρές δυσκολίες, ε, από κρίση. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από μια βόρεια χώρα όπως Σουηδία να ασχοληθεί και με άλλα κλάδους που αφορούν ιδιαίτερα τα μεσογειακά προϊόντα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τεράστιες δυσκολίες στις αγορές. Δεν μπορώ να σιωπήσω για το γεγονός ότι το ο τομέα του ελαιολάδου γνωρίζει σημαντική κρίση, αλλά όπω και τα απορροκυπευτικά. Καλό λοιπόν την Προεδρία να ασχοληθεί παράλληλα με τον γαλακτοκομικό τομέα και με άλλους ε, κλάδους. Και ένα συγκεκριμένο αίτημα τώρα. Δεδομένου του ότι η ανταγωνιστική στρατηγική της ε, κοινωτικής γεωργίας ε, βασίζεται στην διαφοροποίηση και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητα, ε, τι θα πρέπει να γίνει ε, στον τομέα της σήμανσης ε, των ετικετών των τροφίμων, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου ο καταναλωτής να γνωρίζει περί τίνος ακριβώς πρόκειται και να μπορεί να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με την ποιότητα των προϊόντων. Ευχαριστώ κύριε Λαβία, κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την Σουηδική Προεδρία και σαν μέλος από την Ορλανδία ελπίζω ότι όντως θα υπάρξει μια θετική ψήφος στο δημοψήφισμα και ότι θα επικυρωθεί πλέον η σύμβαση. Και ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν πολύ μετά από αυτό. Τέλος πάντων, μιλήσατε για τρόφιμα για όλους. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και κυρίως σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Επίσης ε, μιλήσατε και για την αγορά του γάλακτος και την στη μέσα του γάλακτος και χαίρομαι, όπως είπαν και άλλες ε, συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι, ότι το Συμβούλιο των Υπουργών θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Ε, γιατί πραγματικά είναι επίγον το θέμα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Όλοι όσοι μιλήσαν σήμερα τόνισαν την ανάγκη για επίγουσα δράση. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα, γιατί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τώρα οι γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις ε, είναι σε, κίνδυνο, γιατί μετά την άνοιξη πολλές από αυτές ε, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν, άρα κάτι πρέπει να γίνει βραχυπρόθεσμα και μετά υπάρχει, υπάρχουν και τα μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Μίλησαν γι' αυτό οι άλλοι συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω εγώ. Θα πρέπει να δούμε όλο το σύστημα της αγοράς και να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε έτσι ώστε τα μέσο και μακροπρόθεσμα, μάλλον μέσο και μακροπρόθεσμα να μην δημιουργηθούν ξανά τέτοιου είδους προβλήματα. Ε, υπάρχουν κάποια έλεγχοι αυτή τη στιγμή που δεν λειτουργούν όμως. Ένα αυτό. Α, επίσης αναφερθήκατε και στην κατάληξη του γύρου της Ντόχα. Ε, είπατε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να μην ε, τιμωρηθεί η ευρωπαϊκή γεωργία. Και ελπίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ένα άλλο άλλος τομέας ε, ο οποίος ε, με ενδιαφέρει είναι η μεταφορά των ζώων. Και επειδή ζούμε σε ένα νησί που ζουν πολλά ζώα και τα εξάγουμε στη Γαλλία και στην Ισπανία, το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό για μας και ανησυχούμε. Είπατε στην παρουσίασή σας ότι θα απλουστεύσετε όλους αυτούς τους κανόνες ε, και θα εισάγετε κανόνες που θα είναι εύκολα εφαρμόσιμοι. Ήθελα να ξέρω τι έχετε στο νου σας γι' αυτό. Μετά άλλα δύο θέματα, τα οποία θα ήθελα να επαναλάβω, είπε ο Τζον Νίκολσον για την απλούστευση. Ε, το απλούστευση γίνεται βρισιά, έτσι όπως ε, έχουν γίνει τα πράγματα τώρα και θέλω να ξέρω τι θα είναι διαφορετικό αυτή τη φορά από ό,τι στο παρελθόν. Και κάτι άλλο για την ε, προστασία των εδαφών και την οδηγία θα, υπάρχει, θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Ο κύριος Καλινόνσκι. E, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ευχές που εξέφρασε την άδελφη για την Σουηδική Προεδρία που ανέλαβε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ έχω κατά νου ποικίλα προβλήματα τα οποία πλήττουν τις αγορές μας. Αναφέρθηκε επανειλημμένα ο γαλακτοκομικός τομέας. Η κατάσταση είναι καταστροφική στον κλάδο αυτών. Θα αναφερθώ και σε άλλα θέματα εξίσου σημαντικά. Σημαντικά για τους γεωργούς και όχι μόνο για αυτούς. Παραδείγματος χάρη το ζήτημα των Ε, Σήμερα στην Πολωνία οι τιμές ε, έπεσαν κατά 50-60% σε σχέση με τις τιμές της προηγούμενης χρονιάς, ενώ το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι συμβαίνει με τον κλάδο αυτό, διότι είναι ένα ζήτημα που αφορά και ενδιαφέρει όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια κατάσταση όπου χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, η λήψη κατεπηγών μέτρων ε, παρεμβάσεις οι θα επιτρέψουν στους γεωργούς να αντιδράσουν στην κατάσταση άμεσα. Ε, με τιμές τόσο χαμηλές θα προκαλέσουμε μια άλλη ασφυξία στην αγορά Ε, την κτηνοτροφική ε, και την παραγωγή κτηνοτροφική. Μόρβεϊ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην δραματική και τραγική κατάσταση των αγροτών, κυρίως των μικρών αγροτών, των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στις ε, νέες χώρες, κυρίως στην Ουγγαρία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι αγρότες και γενικά οι χώρες αυτές επηρεάζονται δυσανάλογα από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Γι' αυτό οι αγρότες αυτοί χρειάζονται άμεσα και αποτελεσματικά βήματα έτσι ώστε ε, για να αποφύγουμε την φτώχεια, ε, να αποφύγουμε την ε, πώληση, την εγκατάλειψη των εκμεταλλεύσεων αυτών, προφανώς ε, εμείς έχουμε ιστορικά, ιστορικά έχουμε μειονεκτήματα, ε, δηλαδή όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε και ένα πεβαρημένο παρελθόν. Ε, απ' την άλλη πλευρά όμως γίνανε και κακές ε, και άνδικες ε, συμφωνίες. Εμείς παίρνουμε μικρότερο, ε, μικρότερα ποσά στις επιδοτήσεις από ότι οι αγρότες των παλαιών χωρών και αυτό είναι άδικο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αγρότες ε, των παλαιών χωρών ε, είναι οι εχθροί μας. Όχι, οι εχθροί μας είναι οι πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ, ε, όλοι αυτοί οι οποίοι συμπιέζουν τις τιμές. Και οι αγρότες μας αναγκάστηκαν να αγοράσουν πολύ ακριβά μηχανήματα για να είναι ανταγωνιστικοί. Πήραν δάνεια από τις τράπεζες και Είχαμε και φρικτές κλιματολογικές συνθήκες φέτος, επομένως πραγματικά ζούμε ένα δράμα. Εκατοντάδες ε, αγρότες το φθινόπωρο θα χρεοκοπήσουν. Και αυτό είναι ένας άλλος ε, τομέας, ένας άλλος παράγοντας. Αν, αν υποχρεωθούν ε, να πουλήσουν τις, τα αγροκτήματά τους, θα μεταφερθούν, θα μετακινηθούν στις πόλεις και όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες ε, αγρότες ε, τι θα γίνουνε, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα έχουμε δηλαδή στο κέντρο της Ευρώπης ε, τριτοκοσμικές καταστάσεις από όλο αυτόν τον κόσμο που θα, αναγκαστεί, θα αναγκαστούν να αλλάξουν τον τρόπο να αλλαξουν τροπο ζωη τους, θα μείνουν χωρίς ρίζες, θα εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, στον τόπο τους και θα βρεθούν άστεγοι στις πόλεις. Αυτό είναι δραματική κατάσταση. Όλοι λένε ότι η, πριν από το 2013 δεν μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα των επιδοτήσεων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουμε με τους Ούγγρους ε, αγρότες ή και από τα άλλα νέα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι συναδελφοί από τις νέες χώρες, αλλά σε εμά ε, είναι δραματική η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα σαν δικηγόρος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, με εκπλήσει αυτή η συζήτηση που λαμβάνει χώρα για την διατροφική κυριαρχία, food sovereignty. Είναι μια γενική έννοια Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τρόφιμα, να έχουμε τροφή ποιοτική, δίκαιη και επαρκής. Και θα πρέπει οι τοπικές, οι, τοπι, οι, οι, αγρότες επιτόπου να μπορούν να το, να, θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο και γιατί ε, θα αποφασίσουν, λέτε εσείς. Αυτό είναι ε, το δικαίωμα στην τροφή τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συζήτηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, ε, το social cross compliance είναι μια νέα έννοια. Αυτή την έννοια θα πρέπει να την εισάγουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το social cross compliance. Οι αγρότες οι οποίοι παράγουν δουλειές, θέσεις απασχόλησης δηλαδή, θα πρέπει να έχουν, να παίρνουν περαιτέρω ε, επιδοτήσεις, διότι επιλύουν και κάποια, κάποια προβλήματα ε, οικονομικά και αναλαμβάνουν ε, την ευθύνη να παράγουν θέσεις απασχόλησης και σαν αντάλλαγμα παίρνουν ε, κάποια χρήματα. Ο Γκαρσία Περέσε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Πρώτα απ' όλα διότι τα τη της Προεδρίας θα σημάνουν ότι είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στην σημερινή κατάσταση που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φυσικά λοιπόν και εγώ συμφωνώ με τις ευχές ε, τώρα σήμερα. Μάλλον χθε ρωτήσαμε την Επίτροπε, όπως ε, ρωτάμε και εσάς σήμερα, πάνω σε ζητήματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κλίση στον γαλακτοκομικό τομέα και θα ήθελα να ε, τονίσω την αναγκαιότητα για ύπαρξη περισσότερων κοινοτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κρίση που φυσικά έχει ιδιαιτερότητες σε κάθε μια χώρα, αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκής κρίσης χρειάζεται η λήψη και ευρωπαϊκών μέτρων, διότι τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμόσει μέχρι τώρα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν. Θα θέλω να γνωρίζω λοιπόν ποιε είναι οι προτάσει που θα μπορούσατε να κάνετε από πλευρά Προεδρία. Και μία ερώτηση σχετικά με τις προβλέψεις της Προεδρίας ε, σε θέματα διαφοράς και διαφοροποίησης ε, τιμών. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις ε, τιμές παραγωγού και τις τιμές καταναλωτή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα μας καταδεικνύει ότι πρέπει να θέσουμε σε ε, μηχανισμό κάποιες ε, ενέργειες, μάλλον κάποιες δράσεις. Γνωρίζετε εξάλλου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια, μια βεντάλια και μια, ένας, ένας χώρος ποικίλων καταστάσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας ε, ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν οι μεσονομικέ προοπτικές ε, πάνω στο θέμα αυτό να τροποποιηθούν, να βελτιωθούν, διότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την μοναδική ελπίδα για επιβίωση του κτηνοτροφικού τομέα στην Ευρώπη. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτός από την υποστήριξη που ε, δίνω στον κύριο Νίκολσον για την ρύθμιση απορρίθμιση. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα βιοκαύσιμα, την κλιματική αλλαγή και την ε, επάρκεια ενέργειας. Για την αλλαγή του κλίματος ε, παρακαλώ να παραμείνουμε ρεαλιστές και να μην παρασυρθούμε από τα παχιά λόγια αποτυχημένων Αμερικανών Προέδρων αλλά να παραμείνουμε ριζωμένοι στην πραγματικότητα. Ε, στην Ανατολική Αγγλία από που κατάγουμε ε, ε, πέρσι χιόνισε έξι φορές και όμως με έχουν ζαλίσει με την θέρμανση, υπερθέρμανση του πλανήτη, το global warming. Και επίσης ε, βροχή, βροχοπτώσεις τις οποίες χρειαζόμαστε επιγόντως ε, για στα χωράφια μας και από τις βροχοπτώσεις αυτές δεν είχαμε ανεπάρκεια, ευχαριστημένοι είμαστε. Ας εξετάσουμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή τα επιστημονικά στοιχεία πριν, πριν ακολουθήσουμε ε, ε, άγνωστους και επικίνδυνους δρόμους. Ε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έγινε με τον αυθόδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 67-68 είχαμε μια μεγάλη επιδημία και μάθαμε από τα παθήματά μας. Και είχαμε μια επιτροπή γεωργίας που μας έλεγε σκότωνε και θάψε, σκότωνε και θάψε και το 2001 είχαμε πάλι αυτό ε, και είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έλεγε σκότωνε και κάψε, σκότωνε και κάψε και γεμίσαμε πυρές ε, από σκοτωμένα ζώα ε, με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Γι' αυτό λοιπόν να μάθουμε από τα παθήματα του παρελθόντος. Για τα βιοκαύσιμα ήμουν αρκετά ανόητος και ε, φύτεψα ε, ορισμένα εκτάρια μετά από ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως το οποίο είδα ότι το κόστος, που μου, το κόστος της ενέργειας και η κατανάλωση μάλλον ενέργειας κατά πολύ ξεπέρασε το, όφελος από την καλλιέργεια του, του βιοκαύσιμου. στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αυστηρή ε, νομοθεσία για την χρήση ε, λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων. Ε, Από την άλλη πλευρά θέλουμε βεβαίως να ταΐσουμε όλο τον κόσμο. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτές τις αντιφάσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Τάκεν και ε, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον Προεδρεύοντα ε, του Συμβουλίου. Εγώ είμαι από Δανέζα και έχουμε μια άλλη ε, θέση σε αυτή σε αυτό τον αγροτικό τομέα ο οποίος κατακλείζεται από ενισχύσεις και άλλες στους ε, πράσινους έχουμε συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα και ελπίζω να μας υποστηρίξετε. Έχουμε συμφωνήσει στο εξής, ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα τώρα που μας απειλούν με την επανεθνικοποίηση της γεωργίας. Εκ νέου εθνικοποίηση δεν είναι δυνατό να γίνει. Ο προπολογισμό δεν αντέχει τα καινούργια κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να τα βοηθήσουμε βεβαίως να βρεθούν στην ίδια κατάσταση όπως τα παλαιά μέλη, αλλά κάπου θα, θα, δεν θα αντέξει ο προπολογισμό έχει λυγίσει. Ο Δανός Υπουργός Γεωργίας ε, θα απορρίψει αυτές τις προτάσεις και εμείς ε, οι πράσινοι και εμείς θα απορρίψουμε αυτή την ε, πρόταση και πρέπει και το Συμβούλιο να αντισταθεί. Ξέρω ότι η Επίτροπος είναι εναντίον, αλλά ε, δεν ξέρω τι πιστεύουν οι άλλοι Επίτροποι, τι γίνεται μέσα στην Κομισιό όσον αφορά την επανεθνικοποίηση των ενισχύσεων. Εμείς είμαστε εναντίον και θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Ε, δεν είναι δυνατόν να επαναθνικοποιήσουμε την ε, ΚΑΠ. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημά μου. Ε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ό,τι φορά τις διαπραγματεύσεις που διεξαγόνται με την Ουκρανία. Η χώρα αυτή έχει ένα δυναμικό το οποίο παραμένει αχρησιμοποιητό προς το παρόν στον τομέα της Γεωργίας. Υπάρχουν γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που μεταφέρονται στην περιοχή δημιουργώντας ε, τεράστιες εκμεταλλεύσεις. Μία συμφωνία ελεύθερης ε, αγοράς θα άνοιγε το εμπόριο ανάμεσα στην ε, Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα στρέβλωνε σημαντικά το εμπόριο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι στην Ουκρανία υπάρχουν ε, μια σειρά αριθμίσεων που απέχουν σημαντικά από αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πολύ ευνοϊκό στον τομέα των δημητριακών για τους Ουκρανούς. Ορισμένα κόστη είναι πάρα πολύ χαμηλά διότι έχουν ένα σύστημα διπλής τιμολόγησης για το, στον τομέα της ενέργειας αλλά και πάρα πολλές ζωοτροφές κοστίζουν πολύ λίγο. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αποβαίνουν προς όφελος ε, των ε, παραγωγών της Ουκρανίας αλλά το ίδιο ισχύει και για τον κτηνοτροφικό τομέα όπου δεν προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία των ζώων, την καλή μεταχείρισή τους κλπ. Πολλά μέρη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ουγγαρία γειτονεύουν με την Ουκρανία. Λοιπόν, αν συνεχθεί μια συμφωνία ελεύθερης αγοράς ε, με την Ουκρανία και δεν φροντίσουμε να διασφαλίσουμε κάποιες ε, συνθήκες και την συμμόρφωση των γεωργών και κτηνοτρόφων με, ε, με όσα ισχύουν στην Ευρώπη, τότε καταλαβαίνετε ότι η πολλοί γεωργοί θα μετακινηθούν στην περιοχή αυτή και θα κάνουν την ίδια εργασία με κόστος πολύ χαμηλότερο. Εγώ θα προτείνω κάτι τέτοιο να επιτρέψουμε να συμβεί. Συχλιεύσκη. Μικρόφωνο παρακαλώ. Έχω, έχω. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει οθετήσει μια γνωμοδότηση για την ελεύθερη διανομή τροφίμων στις, στους φτωχότερους πολίτες της Ευρώπης, της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ε, ε, ε, αυτό λοιπόν πρέπει να αποτελεί ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο να ξεκινήσει την εργασία αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει. Η Προεδρία της Τσεχίας δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία από αυτού. Θα αναθεωρήσει το νομοθετικό πλαίσιο η Σουηδική Προεδρία. σε, έναν τόσο, μια τόσο πλούσια ήπειρο είναι απαράδεκτο τόσα εκατομμύρια πολίτες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ε, θα πρέπει επίσης να ανοίξουν οι αγορές Α, η συζήτηση για το άνοιγμα των αγορών από τρίτες χώρε που γίνεται στα πλαίσια του ΠΟΕ, ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας εμεί. Θα επανέλθουμε σε επιδότηση των παραγωγών. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Διαφορετικά ακόμα περισσότεροι παραγωγοί μας θα χρεοκοπήσουν αν ανοίξουν οι αγορέ ε, από προϊόντα από τρίτων χωρών. Ε, ή, ή θα συγχωνευτούν πολλές παραγωγικές μονάδες και θα παρουσιαστεί μια μονοπωλιακή δομή ε, της γεωργίας όπου όλη η, εξουσ... δύναμη θα συγκεντρώνεται σε, σε ορισμένες και λίγες τεράστιες παραγωγικές μονάδες και θα έχουν σβήσει οι μικροί. Äh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και παρακολούθησα ε, με προσοχή την εισήγησή σας. Σε πολλά θέματα συμφωνώ. Έχω ακόμα όμως τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, χάρηκα που αναφέρατε την απογραφειοκρατικοποίηση, δηλαδή τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και ότι θα συμπεριλάβετε αυτό στην ατζέντα σας. Πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία. Είναι, είναι σημαντικό έργο αυτό. Και πιο συγκεκριμένα, με ανησυχεί με, με επειδή αναφέρεται την καμπύλη των αγκουριών και το ποσοστό καμπυ, με ανησυχεί η προστασία των εδαφών. Θα λύσουμε το πρόβλημα της προστασίας των γεωργικών εδαφών ε, στην, ε, στην ευχαίρεια των κρατών μελών ε, ή θα αποφασιστεί κάποιο νομοθετικό πλαίσιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο που πιστεύω θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διοικητικό βάρος. Εγώ θα ήθελα να παραμείνει αυτό στην ευχαίρεια των κρατών μελών. Εν συνεχεία, προκλήσεις λόγω του κλίματος και των κλιματικών αλλαγών Συγχύζουμε κάθε φορά που κατηγορούν τους παραγωγούς ότι ε, η συμβολή τους είναι αρνητική ε, στην προστασία του περιβάλλοντος και ότι συνεχώς ζημιώνουν και βλάπτουν το περιβάλλον. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα επαναξετάσετε την προσφορά και τη συμβολή, τη θετική δηλαδή προσφορά των ε, γεωργών ε, στον αγροτικό τομέα και το ρόλο που παίζουν ε, θετικά στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Τρίτον, έχουμε συζητήσει πολλές φορές την κρίση του γαλακτοκομικού τομέα και σήμερα το πρωί τελευταίο θέμα στην μέση διάταξη της πρωινής συμμεδρίασης ήταν η κατάσταση της αγοράς κρέατος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης όσον αφορά ε, το, τα εισοδήματα των παραγωγών. Λοιπόν, ε, συνδέσατε το θέμα της υγείας των ζώων και της ευζοίας των ζώων, animal health και animal welfare πώς ε, θα χειριστείτε ε, το θέμα της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που πρέπει να εφαρμοστούν στα ζώα ε, έναντι της αύξησης του κόστους παραγωγής. Από τη μία πλευρά θέλουμε σωστά πρότυπα, βεβαίως για να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ευημερία των ζώων, από την άλλη πλευρά όμως δεν θέλουμε τα αύξηση του κόστους και συνεχή επιβάρυνση της τιμής των προϊόντων στην αγορά. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Μάρκο Αντρόμπερ και θα ολοκληρώσω τον κατάλογο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε το θέμα του ΠΟΕ. Αυτό ήταν απόφευκτο, το πράξατε και εσείς Πρόεδρε. Και φράστηκε η ελπίδα ότι θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ. Διαπραγματεύσεις που στο, σε ό,τι αφορά τους ε, μπανανοπαραγωγούς της Ευρώπης ε, είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι βλέπουμε ότι επλήγησαν τα συμφέροντά του και είδαμε ότι έχει υπάρξει μια μείωση των δασμών για τις εισαγωγές ε, μπανάνας. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι η αποψία σχετικά με αυτόν τον πόλεμο της μπανάνας όπως λέγεται και κάτι ακόμα, κατανοώ τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζεται σε αυτή την περίοδο σχετικά με την γεωργία στο σύνολό τη. Το είπαμε και χθε στην ε, κυρία Επίτροπο, το λέμε και σε εσά κύριε Υπουργέ. Πάντως πιστεύω ότι μία από τις δεσμεύσεις θα είναι να διατηρήσουμε την καλλιέργεια μπανάνας και να προστατεύσουμε τους μπανανοπαραγωγούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Εσκύλ, άκουσες ε, μια σειρά ερωτήσεων, έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις και για μια ακόμα φορά σου εύχομαι καλή επιτυχία. Εσκύλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Παύλε και Ευχαριστώ όλους ε, όσοι έθεσαν ερωτήσεις. Ε, εξετίμησα ιδιαίτερα τις ερωτήσεις σας και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να απαντήσω και να σχολιάσω τα σημεία που θέξατε. Ορισμένες ε, ερωτήσεις θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Σε άλλες ερωτήσεις θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ε, όσον αφορά την, τις ετικέτες και την ε, προέλευση, ε, την ενημέρωση του καταναλωτή. Βεβαίως εδώ δεν Θέλουμε να, να, ο καταναλωτής να αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εσφαλμένες πληροφορίες για τη σύσταση από την ετικέτα ή για την προέλευση του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά όμως, ε, είναι γεγονός ότι έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την γεωγραφική προέλευση του προϊόντος σε πολλά τρόφιμα, παραδείγματος χάρη στο βόλιο κρέας, στα ε, νοπά φρούτα και λαχανικά, ήδη αναφέρεται η προέλευση. Και πολλά τρόφιμα σήμερα είναι τρόφιμα τα οποία έχουν συντεθεί από πρώτες ύλες, διαφορετικές πρώτες ύλες και αυτό περιπλέκει την ε, ενημέρωση, τα ενημερωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται. Στο Συμβούλιο λοιπόν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Επίσης, ε, τέθηκε μία συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά, ε, όσον αφορά τις ε, τα, τα, τα, τις πληροφορίες που, δι, δίδονται για κάποιο είδου τυριού. Σε ορισμένα προϊόντα δεν χρειαζόμαστε νέους κανόνες, αλλά οι παραγωγοί θα πρέπει να αναφέρουν ειλικρινά τι περιέχει το τυρί. Ε, εμείς θέλουμε να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό κόστος. Άρα θα πρέπει να ε, ε, δίνουμε βάση στην αρχή της ε, ε, ε, θελούσιας αναφορά στοιχείων. Θα πρέπει να, να είναι λοιπόν ο παραγωγός πρόθυμος χωρίς υποχρέωση νομοθετική να αναφέρει τα στοιχεία, τα συστατικά τα οποία περιέχει το προϊόν του. Βεβαίως ο ΙΕ και ο ΦΑΟ ως ε, υπηρεσία του ΟΗΕ έχει διαπιστώσει ότι θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερες επενδύσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή τροφίμων διεθνώς. Ε, και εδώ και πολύ καιρό αναφέρεται αυτή η ανάγκη περαιτέρω ε, πιστώσεων και, και χρημάτων. Διαπιστώνω τώρα με ικανοποίηση ότι όλο και περισσότερες χώρες αυξάνουν την ε, διεθνή βοήθεια που προσφέρουν ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις του ΟΗΕ. Ε, δηλαδή αυξάνεται η επισητιστική βοήθεια την οποία προσφέρουν πολλά κράτη με στόχο βεβαίως ε, τον σιτισμό των περιοχών που υποφέρουν. για να μπορέσουν να συντηθούν ε, τα εκατομμύρια ανθρώπων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και στα εδάφη, στα γεωργικά δηλαδή, και στους, στην πρώτη ύλη για τις καλλιέργειες και η, επίσης στα, στο δανεισμό. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, γρήγορης ανταπόκρισης σε μικροδάνεια για τους γεωργούς και ε, ιδίως για την αγορά σπόρων, για τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το μικρό παραγωγό, τον τόπιο παραγωγό, ο οποίος θέλει να ε, καλλιεργήσει τα χωράφια του για να πουλήσει ένα μέρος και με το άλλο να στρέψει την οικογένειά του η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρμόδιοι της Γεωργίας από την αρχή του 90 ε, συζητούν τα, γεωργικά θέματα και το μέλλον και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια σχετικά καλή ικανοποιητική θέση όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η Κομισιόν έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να διαπραγματευτεί ε, το, την εντολή του Συμβουλίου, τις εντολές που έχει λάβει από το Συμβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε σωστά διεξαγάγει τις διαβουλεύσεις του γύρου της Ντόχα και βεβαίως μας συμφέρει όλους να ολοκληρωθεί γρήγορα ο γύρος αυτός. Η G20 που συνεδρίασαν πρόσφατα στο Λονδίνο διαπίστωσε ότι ο γύρος, αν ολοκληρωθεί σύντομα γύρω της Ντόχα θα μπορέσει να δώσει ένα καινούριο έναυσμα ε, στη, στο, στο, στις εμπορικές συναλλαγές και στην παγκόσμια οικονομία. Θα μπορέσει να, ε, ε, να τα, ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της ε, στάσιμης οικονομίας, της οικονομικής κρίσης. 150 δις ευρώ ενδέχεται να ε, δημιουργηθεί σαν ε, αν θέλετε, των νέων δραστηριοτήτων. Γι' αυτό ακριβώς ε, θέλουμε όλοι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν της Ντόχα. Για την απλοποίηση τώρα Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στο Συμβούλιο είναι υπέρ ε, της απλοποίησης και ότι θέλουν να προχωρήσουν οι εργασίες. Και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι αυτό το θέλετε κι εσείς. Έτσι λοιπόν ως Προεδρεύων του Συμβουλίου θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ε, μετατρέψω την επιθυμία αυτή σε πραγματικότητα. Ε, είναι μια πολιτική απόφαση διότι την επισημούμε και εμείς αλλά οι καταναλωτές και οι πολίτες μας. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά στην καθημερινή ζωή και των επιχειρήσεων και των παραγωγών. Και γι' αυτό εμείς ως πολιτικοί ε, πρέπει να έχουμε την πολιτική βούληση. Αυτό έχουμε δείξει ότι την έχουμε στο θέμα της απλοποίησης, αλλά πρέπει να δράσουμε και γρήγορα για να προσαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να απλουστευτεί. Εν συνεχεία, είχα πει ε, στην αρχή της ομιλίας μου ότι ε, έχουν παρουσιαστεί προτάσεις 39 συγκεκριμένων απλοποίησεων. Ε, παρουσιάστηκαν τον Μάιο φέτος αυτές τις 39 προτάσεις και η Κομισιόν ε, αναθέσαμε στην Κομισιόν που πληρώνει Συμβουλίου να μας αναφέρει, να μας ε, παρουσιάσει μία εμπεριστατωμένη έκθεση για αυτά τα 39 βήματα απλούστευσης τον Νοέμβριο. Θέμα λοιπόν υψηλής προτεραιότητας. Ε, εν συνεχεία, το ε, επόμενο πακέτο ή το μέλλον της ΚΑΠ και η κρίση του γαλακτοκομικού τομέα. Εδώ διαπιστώνω ότι η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ είχε ξεκινήσει υπό τη Γαλλική Προεδρία και κατά την Προεδρία της Τσεχίας συνεχίστηκαν οι συζητήσεις. Εμείς έχουμε την πρόθεση τον Οκτώβριο να οργανώσουμε μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων για την μέλλον της ΚΑΠ και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα συζητήσουμε τις νέες προκλήσεις, δηλαδή το κλίμα, την ενέργεια, το τομέα της ενέργειας, το γάλα και ε, την ε, ε, κρίση στον τομέα του γάλακτος. Δηλαδή, θα είναι μία σημαντική συμβολή, πιστεύω, η συζήτηση αυτή μετά τη Γαλλική και τη Τσεχική Προεδρία για την έκθεση της Κομισιόν που θα παρουσιαστεί αρχές του καινούριου έτους. Θέλω να δηλώσω σαφώς ότι εγώ υπεραμείνομαι μιας κοινή αγροτικής πολιτικής και θέλω να επιβιώσει βεβαίως το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ΚΑΠ. Όσοι ρωτούν για το μέλλον είναι εν γνώση των λόγων για τον οποίο ε, είναι ε, απολύτως απαραίτητη η ΚΑΠ. Άρα λοιπόν η συζήτηση για το μέλλον είναι μεγάλη σημασίας. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο υπάρχει μεγάλη ένα ευρύτατο ε, κονσένσους για την λήψη μέτρων μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος προϋπολογισμού ε, που θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή γαλακτοπαραγωγή. Και το Συμβουλίο και εγώ ε, βεβαίως ε, θα προωθήσουμε αυτό το θέμα, διότι θα πρέπει να μελετήσουμε τι, τι συμβάλλουν και τι μπορούν να προσφέρουν όλα τα κράτη-μέλη και θα ακούσουμε όλα τα αιτήματα των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Τώρα, από σουδικής πλευράς, όπως σας ήδη είπα, και πιστεύω και υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τους παραγωγούς και ο προϋπολογισμός που έχουμε στα χέρια μας πιστεύω εγώ ότι επαρκεί για να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός μας αρκεί για να καλύψει τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται να ληφθούν ε, για την μετώπιση της οικονομικής κρίσης και ιδίως στον τομέα του γάλακτος. Θα παρουσιάσουμε τις ε, κοινέ θέσεις ε, στον τομέα της γεωργίας αλλά μετά από την μελέτη της έκθεσης της Κομισιόν. είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε την κρίση, μια μεγάλη κρίση σήμερα, πρέπει να την ξεπεράσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα μέσα στα οποία έχουν ε, ήδη ε, χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, εάν θα πρέπει... έχουν τεθεί ερωτήματα μέσα στα, στο πλαίσιο των μέσων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εάν, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να επαναφέρουμε τις επιστροφές εξαγωγών. Δεδομένου ότι ίσως δοθεί έτσι η δυνατότητα ενίσχυσης των φτωχότερων κρατών. γιατί οι φτωχότερες αυτές χώρες είναι σε δυσμενή θέση γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της παραγωγής, της κάλυψης των επιστημιστικών τους αναγών και των εξαγωγών. Η Κομισιόν έχει προτείνει να επεκταθεί η περίοδος ε, παρέμβασης και στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα ληφθεί απόφαση σε αυτή την πρόταση της ε, Κομισιόν και υπάρχει και άλλη πρόταση της Κόμισιον, οι άμεσες πληρωμές. Οι άμεσες πληρωμές στους γεωργούς που θα έπρεπε ήδη να καταβληθούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου για να διευκολυνθεί η λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Άρα λοιπόν καταβολές μέχρι 16 Οκτωβρίου άμεσες πληρωμές. Ε, και η Κομισιόν έχει πει σαφέστατα ότι ζητάει από τις αρχές ανταγωνισμού των διαφόρων κρατών μελών να εξετάσει και να αναλύσει προσεκτικά στις χαμηλές τιμές του γάλακτος και αν αυτές ανταποκρίνονται και σε χαμηλότερες τιμές ε, για τους καταναλωτές. 39% στη Σουηδία έχει μειωθεί η τιμή του γάλακτος. Αλλά για τον καταναλωτή έχει μειωθεί το γάλα μόνο 2%. Οι αρχές ανταγωνισμού λοιπόν σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάσουν λεπτομερώς αυτή την κατάσταση, αυτά τα γεγονότα και να δουν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Όσον αφορά το σύστημα ποσοστώσεων, και για την κατάργηση των ποσοστώσεων στο μέλλον σας παραπέμπω στη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το καλοκαίρι. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι τα συμπεράσματα που έγιναν μετά από τον έλεγχο υγείας ισχύουν όπως έχουν ληφθεί. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα διότι σήμερα υπάρχουν ποσοστώσεις και αυτές οι ποσοστώσεις δεν έχουν αυξηθεί. Παρόλα αυτά έχουμε ε, τιμές παραγωγής που έχουν υποχωρήσει σημαντικότατα. Άρα, γιατί έχουμε ποσοστώσεις, γιατί υπάρχουν οι ποσοστώσεις, δεν έχουν βοηθήσει διόλου τον Ευρωπαίο γαλακτοπαραγωγό, ενώ υποτίθεται ότι αυτό ήταν ο στόχος τους. Γι' αυτό οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν διαπιστώσει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα συμπεράσματα του health check, του ελέγχου υγείας δηλαδή που έγινε. Ε, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ε, ενισχύσεων για τους ε, Ευρωπαίους γεωργούς. Τα επίπεδα τα οποία ισχύουν τώρα ορίστηκαν μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκαναν τα διάφορα κράτη-μέλη με την Ένωση. Μετά το 2013, κατά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να προσαρμοστούν έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή κατανομή από τα ταμεία ε, μέσα στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων που δίδονται. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, περνάω στο θέμα των μεταλλαγμένων. Αυτό είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργήσει, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε πολλά για να μην πω σε όλα τα θεσμικά όργανα της κοινότητας. Και με τους εμπορικούς μας εταίρους ε, έχει, μας έχει προκαλέσει συζητήσεις. Λοιπόν, υπάρχει από τη μία πλευρά οι σπόροι που προέρχονται από μεταλλαγμένα και, τα, και οι οποίοι καλλιεργούνται και δεύτερον οι η σύνθεση, η σύσταση των προϊόντων που περιέχουν μεταλλαγμένα. Για το πρώτο θέμα της καλλιέργειας δεν έχω εγώ καμία θέμα, δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Ο Υπουργό Περιβάλλοντος ασχολείται. Για τα άλλα όμως, για τη σύνθεση των προϊόντων, σύσταση των προϊόντων, ε, εκεί έχω αρμοδιότητα. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είχαμε πει, είχαμε αποφασίσει ότι ούτως ή άλλως ε, εμείς έχουμε μια αυστηρή νομοθεσία και ναι μεν έχουμε προχωρήσει και έχουμε μια πολύ προωθημένη νομοθεσία με την πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας στην εποχή αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή. Από την άλλη πλευρά, όταν παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα επιστημονικά δεδομένα. Η Κομισιό ε, υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει στο Συμβούλιο μία έκθεση. Τη Δευτέρα κιόλας, τώρα, το Σεπτέμβριο και προφανώς θα μπούμε σε λεπτομέρειες στην συζήτηση, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διιστάμενες απόψεις και ίσως η Κομισιό μπορεί να υποβάλει εκ των ημετά ε, και κάποια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτόν τον τρόπο για να λύσουμε το πρόβλημα των μεταλλαγμένων. Τώρα, για τα άλλα θέματα, το ελαιόλαδο. Σημείωσα την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαρθρωτικών της μέτρων δίνει ενίσχυση στο ελαιόλαδο και με την στήριξη των τιμών και με την παρέμβαση για τα δημητριακά. Υπάρχει μια διακύμανση των τιμών. Και η Κομισιό διαχειρίζεται τα προβλήματα αυτά. Ούτως ή άλλως δεν είναι το Συμβούλιο αρμόδιο. Τώρα όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων. Περιμένουμε μια έκθεση από πλευράς της Κομισιόν. Δεν ξέρω πότε θα υποβληθεί η έκθεση αυτή. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας απαντήσει για το θέμα αυτό. Προφανώς εάν η πρόταση αυτή υποβληθεί κατά διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα διότι ακόμα δεν την έχουμε πάρει την έκθεση αυτή. Επομένως Προφανώ δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Τώρα, οι, οι, που δίδονται σε αυτούς που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, σε λιγότερο ευνοϊκή θέση στην κοινότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποστήριξη σε επίπεδο συμβουλίου για τέτοιου είδου πρόταση. Εάν η Κομισιόν τώρα ε, υποβάλει μια αναθεωρημένη πρόταση, η Προεδρία, εγώ δηλαδή, θα προσπαθήσουμε όλες αυτές οι πτυχές να ε, προχωρήσουν λαμβάνοντας υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών. Μέχρι στιγμής όμως το θέμα έχει, είναι μπλοκαρισμένο. Η Ουκρανία. Κατά την άποψή μας, το εμπόριο δημιουργεί ευημερία. Εγώ ε, προέρχομαι από μια χώρα που ε, έχει πολλές εμπορικές συναλλαγές και περάσαμε από το στάδιο μιας φτωχής χώρας ε, στο στάδιο μιας πλούσιας χώρας. Και βλέπουμε, έχω δει δηλαδή πώς, μπορούμε, πώς μπορεί μια φτωχή χώρα να γίνει πλούσια και πιστεύω ότι η Ουκρανία έχει ένα μέλλον μπροστά της. Βέβαια, στην Ευρώπη έχουμε μια παραγωγή ψηλή τεχνολογίας. Οι αγρότες μα είναι καλά καταρτισμένοι. Έχουμε προϊόντα τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε σε καταναλωτές που έχουν ένα υψηλό επίπεδο, αν θέλετε, μια ποιότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ε, όταν συνάπτουμε οποιοδήποτε συμφωνία με την Ουκρανία. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τις άλλες χώρες με τις οποίες συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίες. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των ζώων. Αυτά είναι προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά. Τα θεωρώ δηλαδή και εγώ πολύ, πολύ σημαντικά. Και είναι πολύ σημαντικά και για τους ε, καταναλωτές, ε, τους Ευρωπαίους. Και πολύ συχνά το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τις απόψεις αυτές, ότι τα προβλήματα αυτά είναι σημαντικά δηλαδή ενώ. Αυτό φαίνεται και από το πώς εξετάζει το Κοινοβούλιο τα διαφό τις διάφορες προτάσεις. Ως Σουηδός υπουργό πιστεύω ότι τα υψηλά στάνταρ τα οποία ισχύουν στην Ευρώπη είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό και πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και οι, οι, οι, οι αγρότες μας έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως έχω πει και στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω και τώρα, σαν παλιός αγρότης κι εγώ, ότι τα υγιή ζώα δίνουν μια καλύτερη παραγωγή. Οι χείροι, α πούμε, όταν είναι υγιεί, όχι απλώ μεγαλώνουν καλά, δίνουν και καλύτερα προϊόντα. Α αφήσουμε του χείρου τώρα και προσχωρήσουμε στι μπανάνε. Οι μπανάνες είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Συμμετέχουν πολλοί. Υπάρχουν πολλοί ε, εμπλεκόμενοι εδώ, αν θέλετε. Οι χώρες Λατινικής Αμερικής, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το καθεστώς εισαγωγής των προϊόντων αυτών αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στον ΠΟΕ. Και το καθεστώς το καθεστώς εισαγωγή των μπανανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κριθεί πάρα πολλές φορές ασυμβίβαστο με, την, ε, με τους κανόνες του ΠΟΕ. Εμείς λέμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σεβόμαστε τους κανόνες. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σεβαστούμε τους κανόνες τους οποίους συνεισφέραμε να υιοθετηθούν. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Πάολο, ευχαριστώ και όλους τους ε, βουλευτές. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το απόγευμά μου αυτό και ελπίζω θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα ότι η συναπόφαση έχει αρχίσει να λειτουργεί. Ήδη το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο δουλεύουν μαζί. Ένα λεπτό μόνο διάλειμμα για να χαιρετήσω τον φίλο και συνάδελφο που ήρθε εδώ